the camera uh-huh. will take me and you what to... So, uh, dear colleagues, uh, good morning. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος. Καλώς ορίσατε. Ξαναρχόμαστε εδώ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μετά τις διακοπές. Ελπίζω ότι ξεκουραστήκατε στις διακοπές όλοι σας. Και τώρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζεστό μάλλον, φθινόπωρο, ζεστό τέλο πάντων σε κάποια κρατημέλη, καυτό, καυτό σε κάποια κρατημέλη που θα έχουν εκλογέ και άλλες εξελίξεις. Οπότε ξεκινούμε τη σημερινή μα συνεδρίαση. Θα προεδρεύσω αντί του κυρίου Λάγκε, του πρόεδρου μα. Το πρώτο μας σημείο στη μεσαία διάταξη είναι η έγκριση της ε, την έγκριση αυτή. Οπότε τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή. Έχουμε το σημείο υπάρχει μόνο αυτό. και το οποίο θα το συζητήσουμε πριν την κοινή συζήτηση το 6 δηλαδή και το 7 δηλαδή την έκθεση για το Καζαχστάν. Αν δεν έχετε κάποια ένσταση να εγκρίνουμε τη μέση διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ένταση, Επομένω, εγκρίνεται η μέση διάταξή μα με αυτή τη μεταβολή. Τώρα πάμε στο δεύτερο σημείο που είναι η έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεις 19 και 20 Ιουνίου αλλά και 10 και 11 Ιουλίου ενιστότος έτους αν δεν ε, διατυπωθεί κάποια ένσταση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά θα είναι εγκεκριμένα. Πάμε τώρα στο σημείο 3 της που είναι η ανακοινώση του Προέδρου για τις αποφάσεις των συντονιστών. Οι αποφάσεις των συντονιστών κατά τη συνάντηση της 19ης Ιουνίου αλλά και 10ης Ιουλίου περιέχονται στα πρακτικά οπότε και αυτές οι αποφάσεις εγκρίνονται αφού δεν διατυπωθεί κάποια ένσταση μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Και σας ευχαριστώ. Ανακοίνωση του Προέδρου, το σημείο 4, ως συνήθως, θα μεταδίδεται στο ίντερνετ η συνεδρίασή μας και έχουμε και διερμηνία και, και οπότε να καλημερίσουμε όλους μας τους θεατές και ακροατές του διαδικτύου και για να διευκολύνουμε το έργο των ε, διερμηνέων θα πρέπει να μιλάμε σε, με κάποια λογική ταχύτητα. Και τώρα η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες όσον αφορά τις συμφωνίες εμπορικού χαρακτήρα με δηλαδή και Αυστραλία δεν έχουν ανακοινωθεί στις 11 Ιουλίου στην τελευταία μας συνάντηση. Πάντως θα συζητήσουμε του κυρίου Κάσπαρη όσον αφορά τι συστάσει για αυτέ τι διαπραγματεύσει με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Πάντω ε, αυτή η ημερομηνία θα είναι 29 στι 6 η ώρα. Τώρα κάποια νέα εμπορικού χαρακτήρα. Η γενικό χαρακτήρα περιοχή ελευθέρου εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανίας ε, τώρα έχει ανοίξει πλήρω την 1η από το 2016 και στη, την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 έχουμε την Συμφωνία σύνδεση. και οι εσωτερικέ διαδικασίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώθηκαν στι 11 Ιουλίου. Και είπαμε ότι έχουμε τώρα στις 17 Ιουλίου την έγκριση από το Συμβούλιο τις θέσεις του Κοινοβουλίου στην πρώτη ε, ανάγνωση. Πρόκειται να γίνει υπογραφή της ε, συμφωνίας για αυτά τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα στην επόμενη σύνοδο στο Στρασβούργο και μόλις γίνει δημοσίευση θα τεθεί σε εφαρμογή. Επίσης έχουμε τώρα ενημέρωση όσον αφορά το πώς πάντα πράγματα όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις του τεμέρους διαλόγου. Είναι μια τέτοια συνάντηση από την τελευταία μας, δική μας συνάντηση στις 12 Ιουλίου και έχουμε τώρα την πρόταση όσον αφορά τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού ε, για το anti Είναι ο Σολτόρη Τσίκου ο εισηγητή και η δεύτερη συνάντηση πρέπει να γίνει αύριο, 31η Αυγούστου. Don't see the rapporteur, so I'm, uh, uh... Αλλά δεν βλέπω να έχει έρθει εδώ ο εισηγητή μα. Οπότε σα υπενθυμίζω ότι ο στόχο αυτή τη πρόταση είναι να θεσπιστεί μια τέτοια νέα μεθοδολογία ούτω ώστε να καλύψουμε ε, το ντάμπινγκ των εισαγωγών που έρχονται σε κάποιε χώρε που υπάρχουν κάποιε τρευλώσει και ε, επίση έχουμε την έκθεση που εγκρίθηκε τον Ιούνιο και η πρώτη τριμή συνάντηση θα γίνει στις 12, έγινε στι 12 Εβδόμου και ήταν πάρα πολύ επικοδομητική, είχε τα βασικά σημεία τη ε, πρόταση και όλα αυτά πρέπει να, να συζητηθούν και πάλι στην αυριανή δεύτερη συνάντηση και πρόκειται ο εισηγητή μα κάποια στιγμή να μα ενημερώσει. Οπότε, όπως θυμάστε, είπαμε ότι θα γίνει αλλαγή μέσα σε διάταξη και γι' αυτό τώρα πάμε στο σημείο 8 το οποίο είναι οι κανόνε και οι αρχέ σχετικά με του τρόπου ελέγχου από τα κράτη-μέλη για την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Συντάκτη είναι ο Βιμ Φαντεκάμπ. Έγινε τώρα η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την γνωμοδότησή μα όσον αφορά την νομοθετική πρόταση που διέπεται από τις διατάξεις της Επιτροπολογίας και ε, η Νομική Επιτροπή είναι κυρίως αρμόδια οπότε και τώρα θα δώσουμε τη σκητάλη στον εισηγητή μας τον Βιμ Φαντεκάμπ για να κάνει την εισήγηση του Συνάδελφοι, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω Ελπίζω ότι γυρίζετε υγιείς και ξεκούραστοι. Ε, θα έλεγα να ελπίζω ότι επιβιώσατε τον διακοπών, αλλά θα ήταν πολύ αρνητικό. Ελπίζω τελο πάντων να τις χαρήκατε. Είμαστε φαντάζομαι όλοι έτοιμοι να ξαναγυρίσουμε στα καθήκοντά μας. Η τροπολογία επί του κανονισμού επιτροπολογίας ε, δεν είναι από τα πιο ελκυστικά θέματα δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ε, προκαλέσει τους δημοσιογράφους ή θα τους έλξει ή θα τους ε, εμπνεύσει να γράψουν. Όμως ε, είναι πολιτικά ιδιαίτερα ευαίσθητο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ιδιαίτερα τεχνικό θέμα, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα εφαρμοστικά. Πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και παλιότερα. Ε, Είχαμε περιπτώσεις όπου η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβουλίο είχαν δεχτεί προτάσεις ε, της Κομισιόν, ε, αλλά που η εφαρμογή τους τελικά δεν επετεύχθη από τα κράτη-μέλη. Ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης πέρσι είχε πει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εμάς εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Εργαζόμαστε επί σοβαρών ευαίσθητων θεμάτων. Για παράδειγμα είχαμε τη ΣΕΤΑ τελευταία, αλλά είχαμε και ορισμένα τμήματα της TTIP, πολύ ευαίσθητα. Αν λοιπόν παίρνουμε αποφάσει κάποιε χρονικέ στιγμέ οι οποίε δεν εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη αργότερα ή αν τελικά τα κράτη, ή αν τα κράτη-μέλη ακολουθούν μια πολύ ουδέτερη στάση, αυτό πλήττει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρόφιμα, γεωργία, εμπόριο, ε, τελωνία, όλα αυτά είναι ευαίσθητα ζητήματα, είναι ζητήματα που έχουν ευαίσθητε πτυχές. Εγώ βλέπω θετικά αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Δεν έχω ακόμα μιλήσει με τους κοιόδης ηγητές, αλλά πιστεύω θα ήταν καλό να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος Επιτροπής και άλλοι επίτροποι, να τα λάβουμε υπόψη μας, διότι οι τροποποίησεις του κανονισμού επιτροπολογίας πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Δεν πρόκειται για μια εκβάθρον ανανέωση του κανονισμού, πρόκειται για μια βελτιστοποίηση ορισμένων σημείων του, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη ε, θα ε, αναφέρουν, θα υποβάλουν εκθέσεις για τις ε, αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτές εφαρμόστηκαν. Έχω βέβαια και εγώ έχω μερικές ερωτήσεις και απορίες αν η απόφαση φτάσει στην ε, Επιτροπή Προσφυγών για δεύτερη φορά. Αναφέρεται από την Κομισιόν ότι θα πρέπει το θέμα να παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή σε κάποια επιτροπή του Συμβουλίου τουλάχιστον. Μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό η Κομισιόν. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να, ξανα, ε, θα πρέπει να δημοσιεύονται οι ψήφοι το πώς ψήφισε κάθε ε, μέλος της Επιτροπής ε, Προσφυγών. Ε, αυτό για να οθηθούν τα κρατημένα, να λαμβάνουν θέση. Μπορεί να μου το επιβεβαιώσει και αυτό η Κομισιόν. Μετά, η, ένα από τα κρατη η Τσεχική Δημοκρατία, νομίζω, ρώτησε γιατί δεν έχει γίνει μελέτη επιπτώσεων, η αξιολόγηση επιπτώσεων. Προσωπικά πιστεύω δεν, δεν έχει σημασία. Αλλά ας τεθεί και αυτό ε, αυτό το ερώτημα εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Είναι ερώτημα του Κοινοβουλίου της Τσεχίας. Το ζήτημα αυτό είναι πολιτικά ευαίσθητο και συμφωνώ με την Κομισιόν, είναι απολύτως απαραίτητο να γίνουν αυτές οι αλλαγές γιατί τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να αποφεύγουν τις ε, ε υποχρεώσεις, τις θεσμικές υποχρεώσεις θα συνεργαστούμε την Κομισιόν για να καταλήξουμε κάπου πολύ σύντομα. Κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές ότι ε, έχουμε περιόριστο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά σίγουρα πολλές φορές μπορούμε να επιταχύνουμε. Ευχαριστώ. Uh, thank you, uh, uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιγητά και επειδή τώρα είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν στα μέλη της Επιτροπής μας. Έχουμε λοιπόν δύο συναδέλφους από την Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κλάους. Παρακαλώ κύριε Κλάους. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Βαντεκάμπ ε, για τις ε, θετικές του παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση Επιτροπής. Ο κύριος Βαντεκάμπ πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του κυρίου Γιούγκα πριν από ένα ακριβώ χρόνο στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ένωση. Τότε παρουσίασε την πρόταση της Επιτροπής. Βεβαίω, αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθούμε να υπερκεράσουμε την διαδικασία της επιτροπολογίας, αλλά σημαίνει ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως είπε και ο κύριος Βαντεκάμπ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι γενικά το θέμα της επιτροπολογίας λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Να αναφέρω και ένα στοιχείο, περίπου 1500 εφαρμοστικά μέτρα εγκρίνονται κάθε χρόνο και το 98% αυτών την χάνουν ε, θετικής ε, προσέγγισης ε, στις επιτροπές της Επιτροπολογίας. Οι επιτροπές δεν τοποθετούνται σχεδόν ποτέ αρνητικά έχουμε ένα 2% περίπου, ε, χωρίς ε, άποψη αποχή δηλαδή, στο αποτέλεσμα ψηφοφοριών στις επιτροπές. Άρα δηλαδή μετά την ε, ψηφοφορία δεν προκύπτει ούτε ειδική πλειοψηφία, ούτε αρνητική στάση κατά των εφαρμοστικών μέτρων. Αυτό λοιπόν το θέμα της μη τοποθέτησης, της αποχής, αυτό θέλει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν καταστάσεις όπου, όπως προβλέπει και ο κανονισμός, αν δούμε λιγάκι την προστασία της ε, υγείας ε, ανθρώπων, ε, εμβιονόντων, ανθρώπων και φυτών, αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και ακριβώς αυτό έχουμε ακριβώς αυτό το 2%, όπου δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως τοποθέτηση και παίζει ρόλο. Και σε αυτό ακριβώς το θέμα τα κράτη-μέλη, πολύ περισσότερο από ό,τι θα επιθυμούσαμε, τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να τοποθετηθούν με σαφήνεια, δηλαδή είτε να στηρίξουν ε, το νομοθετικό μέτρο, είτε να το ε, καταψηφίσουν. Και τι κάνουν, αφήνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει για το τι πρέπει να γίνει. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιο, κάποια διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσει, δηλαδή αν θα προχωρήσει με το μέτρο ή όχι, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο ευαίσθητο θέμα ε, της γλυφοσάτης ή των μεταλλαγμένων οργανισμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διακριτική ευχαίρεια, αλλά είναι υποχρεωμένη να λάβει απόφαση μετά από αίτημα αδειοδότησης ενός προϊόντος σε μια ουσία, εφόσον αυτό το αίτημα κατατεθεί από έναν ε, παραγωγό. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η Επιτροπή δεν μπορεί να πει ότι δεν αποφασίζουμε, είναι υποχρεωμένη να αποφασίσει. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, πέρυσι ο κύριος Γιούγκερ στην έκθεσή του για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση από τα κράτη-μέλη. Όταν δηλαδή υπάρχουν ευαίσθητο θέμα να ε, ρίχνει την καυτή πατάτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ξεκινάνε δύσκολες συζητήσεις ε, στα μέσα ενημέρωσης. Άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευαισθητοποιήσει τα κράτη-μέλη, να τοποθετούνται με σαφήνεια σε προτινόμενα μέτρα και η Επιτροπή μετά να λέει ναι ή όχι και με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί ο στόχος ε, λήψης μέτρων. Το πρώτο μέτρο είναι να αλλάξουν οι κανονισμοί ψηφοφορίας για την επιτροπολογία. Δηλαδή, θα μετρώνται, προσμετρώνται μόνο αυτές οι ψήφοι όπου καταρχήν τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην ψηφορία και κατά δεύτερον ψηφίζουν υπέρ κατά. Δηλαδή ε, εκεί όπου τα κράτη-μέλη δεν είναι παρόντα ή δηλώνουν αποχή, αυτές οι ψήφοι δεν προσμετρώνται στην ψηφοφορία. Η δεύτερη πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα να Συγγνώμη, κάτι πράγμα δεν έχω πει με εννοία. Ότι όλες αυτές οι προτινόμενες αλλαγές αφορούν μόνο την Επιτροπή και την κατάσταση μετά την ε, ψηφοφορία στις επιτροπές. Και στην περίπτωση αυτή το όλο θέμα παραπέμπεται στην επόμενη επιτροπή. Σε αυτή λοιπόν τη φάση γίνεται λόγος για τις αλλαγές που μπορούν να προκύψουν. Είπα ότι θα γίνουν αλλαγές, προτείνουμε αλλαγές ε, στην, ε, στις ψήφους που θα προσμετρώνται στην ε, δεύτερη επιτροπή, μετά στις δυνατότητες που θα μπορεί κανείς ε, να τοποθετηθεί μετά το αποτέλεσμα της δεύτερης επιτροπής, να πάει δηλαδή το θέμα ακόμα πιο πάνω στο Συμβούλιο των Υπουργών, με άλλα λόγια, η δεύτερη αυτή επιτροπή, όπου υπάρχει προσφυγή, αυτή παίζει κάποιο ρόλο, αλλά προβλέπεται ότι τελικά οι υπουργοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να αναζητήσουν μία λύση. Ένα τρίτο στοιχείο, τρίτη προτινόμενη αλλαγή, είναι να υπάρχει δυνατότητα το θέμα να παραπέμπεται στο Συμβούλιο. Δηλαδή, να φεύγει από την Επιτροπή Προσφυγής, να γίνεται πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο και να επανέλθει το θέμα αν δεν αποφασίζει το Συμβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο δεν έχει θεσμικό ρόλο στην Επιτροπολογία το τέταρτο στοιχείο της πρότασής μας και το τελευταίο είναι ότι επιθυμούμε να υπάρχει διαφάνεια στην ε, ψηφοφορία και στην ψήφο των κρατών μελών. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε διαφάνεια μόνο όσον αφορά το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας. Αλλά δεν έχουμε διαφάνεια, δεν ξέρουμε ε, το πώς ψηφίζει ένα κράτος μέλος, αν υπερψηφίζει, καταψηφίζει, δηλώνει αποχή. Άρα δηλαδή και αυτό το στοιχείο είναι καινούριο. Αυτές τις τέσσερις αλλαγές ε, προτείνουμε. Σας λέω, δεν είναι ότι γίνεται επανάσταση στον κανονισμό περί επιτροπολογίας, απλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα σε ε, θέματα που έχουν κάποια πολιτική ευαισθησία και νομίζω ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και αυτός μπορεί να σας δώσει πληροφορίες από αυτό το πρίσμα και θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Πρόεδρος, ε, και εγώ αυτό ήθελα να πω ότι πρέπει να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Νταπίλ σχετικά με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Να σας ε, εκθέσω κι εγώ ποια είναι η αξιολόγηση από τη δική μας πλευρά αυτής της πρότασης. Στο, στον τομέα του, της εμπορικής πολιτικής η επιτροπολογία εφαρμόζεται στην λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2014 η υιοθέτηση τέτοιων μέτρων, εμπορικών μέτρων άμυνας, ήταν εκτός, της επιτροπής, εκτός των κανόνων της επιτροπολογίας. Αυτό όμως άλλαξε το Φεβρουάριο του 2014. Είναι κάτι σχετικά καινούριο λοιπόν. Εμείς υποκείμεθα σε δύο τύπους διαδικασιών, την συμβουλευτική διαδικασία και την διαδικασία εξέτασης, η οποία εφαρμόζεται στην υιοθέτηση οριστικών μέτρων εμπορικής άμυνας, για παράδειγμα ή εναντίον ε, μέτρων ε, κατά παράνομων ε, ε, χρηματοδοτήσεων. Ε, η επιτροπολογία εφαρμόζεται με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, τις οποίες θα σας αναφέρω, κατά την ε, στην Επιτροπή Εξέτασης η ψηφοφορία γίνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία και εκεί έχουμε διάφορα σενάρια. Για παράδειγμα, μπορεί να δοθεί θετική γνωμοδότηση με ειδική πλειοψηφία από την Επιτροπή εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν θα πρέπει να υιοθετήσει την πρότασή της τελικά, την πρόταση που είχε υποβάλει στην Επιτροπή. Ένα άλλο σενάριο είναι να μην, η απουσία γνώμης, δηλαδή να μην σχηματιστεί η ειδική πλειοψηφία, να μην εξασφαλιστεί η ειδική πλειοψηφία. Εδώ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες γιατί έχουμε δύο υποσενάρια. Για παρα... Ε, πρώτον, απουσία γνώμης αλλά και απουσία ε, σχετικής Σε αυτή την περίπτωση ο κανονισμός αναφέρει ότι η Κομισιόν μπορεί να υιοθετήσει την πρόταση που είχε υποβάλει. Υπάρχει όμως και το άλλο υποσενάριο, να έχουμε απουσία γνώμης αλλά εξασφάλιση της σχετικής πλειοψηφίας κατά της πρότασης Κομισιόν. Σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκινήσει την ε, προσφυγή στην Επιτροπή Προσφυγών. Αυτό είναι η ευθύνη ιδιαιτερότητα στον τομέα του εμπορίου. Στην, Επιτροπή, στην διαδικασία εξέτασης, αν το αποτέλεσμα είναι αρνητική γνωμοδότηση και πάλι πρέπει να πάμε στην Επιτροπή Προσφυγών. Όταν δηλαδή εξασφαλιστεί η δική πλειοψηφία κατά. Από το Φεβρουάριο 2014 και μετά η κατάσταση είναι ως εξής. Η διαδικασία προσφυγής ε, έχει πυροδοτηθεί, έχει χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά παρόλο ότι ε, πολλά θέματα έχουν περάσει από την διαδικασία εξέτασης. Εκεί σχεδόν πάντα έχουμε ή θετική γνώμη ή απουσία γνώμης, οπότε η Κομισιόν συνήθως υιοθετεί την πρότασή της. Η μόνη περίπτωση χρήσης της ε, διαδικασίας προσφυγών ήταν το Φεβρουάριο 2017 πρόσφατα ε, στην περίπτωση των ηλιακών πάνελ που ήταν λίγο πιο περίπλοκη από άλλες περιπτώσεις. Η δική μας γνώμη λοιπόν είναι ότι δεδομένων, των, δεδομένων του πολύ μικρού αριθμού προσφυγών που είχαμε στο δικό μας τομέα, η πρόταση αυτή θα έχει ελάχιστο ασήμαντος μηδαμινό αποτέλεσμα στον τομέα μας, ε, στον κλάδο μας. Δηλαδή η αλλαγή στον, στους κανόνες πληροφορίας στην Επιτροπή Προσφυγών θα έχει πολύ μικρές συνέπειες. Ε, η δε πρόταση για παραπομπή στο Συμβούλιο ε, θα ήθελα να σας πω ότι οι δικές μας περιπτώσεις ε, και οι δικές μας αξιολογίες στον τομέα του εξωτερικού μπορεί βασίζονται σε τεχνικούς και νομικούς πολύ σαφείς τεχνικούς και νομικούς παράγοντες και κριτήρια και επίσης έχουμε και συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Οπότε η παραπομπή σε υψηλότερο επίπεδο στους υπουργούς, κατ' εξαίρεση βέβαια, ε, στην περίπτωση που εμφανίζεται απουσία γνώμη στην Επιτροπή, θα πρέπει να σταθμιστεί από τις ανάγκες να τηρηθούν οι ε, εκ του νόμου προερχόμενες ε, προθεσμίες. Οπότε και πάλι ε, μετριάζονται ακόμα περισσότερο οι πτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η πρόταση στο δικό μας τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για τα όσα μας εκθέσατε. Και τώρα στρεφόμεθα προς τους συναδέλφους, έχουμε τους κοιόδης εισηγητές, αλλά και τους άλλους συναδέλφους, πρώτα-πρώτα από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Εμμανουέλ Μορέρα είναι σκιώδης ε, αλλά θα μιλήσω ε, ανταυτού γιατί δεν μπόρεσε να παραστεί και συμφωνεί ο σκιώδης λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αποδείχθηκε ότι δεν αποδίδει η Επιτροπολή για τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν ε, υπάρχει πολιτική λογοδοσία και γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί θεμητέ επικρίσεις γιατί το σύστημα δεν ε, δείχνεται από διαφάνεια. Οπότε θα πρέπει να δούμε στην Επιτροπή τι γίνεται με τα θέματα περιβάλλοντος και υγείας, ούτε εκεί υπήρξε διαφάνεια και επίσης αυτό προκύπτει και στα θέματα εμπορικής πολιτικής και θυμόμαστε όλοι τι έγινε όταν είχαμε στην Επιτροπή τους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Δεν είχαμε την ευρετή απαρτία για να εγκρίνουμε ε, τα ε, μέτρα αντιντάμπινγκ για τα ηλιακά πάνελ. Οπότε ε, γι' αυτό και έλαβε η Επιτροπή την ευθύνη του να αποφασίσει κατά πόσο θα γίνει η παράταση της ισχύω των μέτρων και επομένως έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο υποσχόμαστε, αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί και είπαμε ο κύριος Μωράς θα συμφωνήσει να αλλάξουν οι κανόνες για την ε, ψηφοφορία και έτσι τα κράτη-μέλη να τοποθετηθούν για όλα τα θέματα. Να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τους κανόνες της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο και να αποφασίσει το Συμβούλιο και όχι οι τεχνοκράτες. Όμως λέει ο εισηγητής μας ότι με αυτές τις αλλαγές ε, δεν τρίτη υποσχέσει το του τη επιτροπή ότι θα πρέπει να έχει πιο πολιτικό χαρακτήρα η δράση τη Επιτροπής. Θα πρέπει επομένω κάτι να γίνει για τι θεσμικέ ρυθμίσει, να έχει πιο αποφασιστικό ρόλο το Κοινοβούλιο. Θα συνεργαστούμε πάντω με τον εισηγητή και του άλλου και του και ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να είναι καρποφόρα. Σα ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Τώρα, το ECR και οι Άλντε ε, έχουν σειρά, αλλά δεν βλέπω να παρίστανται. Γκουε, οι πράσινοι, ούτε οι εκείνοι θέλουν να λάβουν το λόγο, ούτε το EFDD. Οπότε, για να το με τώρα, οι υπόλοιποι συνάδελφοι της Επιτροπής, όσοι έχουν στήσει τον ε, λόγο, κυρία Ρόβολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν στα Ολλανδικά ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε, γιατί πράγματι είναι ένα θέμα που δεν αρέσει σε κανένα. Και δεν αρέσει γιατί ε, δεν ε, συνοδεύεται ε, με θετική απήχηση, θα έλεγα. Και τώρα, κάποιες δικές μου σκέψεις όσον αφορά τη συζήτηση για τη κατεξοδότηση πράξης, για την επιτροπολογία, τον έλεγχο της επιτροπολογίας, ε, ε, τον έλεγχο των επιπτώσεων. Αυτά γίνονται εδώ και χρόνια. Και στη τελική ανάλυση τίποτα δεν αλλάζει. Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Τώρα το σύγκρουση μπορεί να είναι λίγο πολύ, ας το πούμε, αντιπαράθεση αν θέλετε. Υπάρχει κάποια διαφωνία ανάμεσα στους ε, θεσμού για τι αρμοδιότητες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι τα κράτη-μέλη μοιάζουν να μην κατανοούν ότι τελικά οι δικοί τους υπουργοί είναι εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο Συμβούλιο. Και τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Δίνουν την εντύπωση ότι ό,τι αποφασίζεται στις Βρυξέλλες δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εγώ χαίρομαι που επιτέλους, θέλω να ελπίζω, επιτέλους θα κατορθώσουμε να γνωστοποιείται το, η συμμετοχή στην ψηφοφορία. Νομίζω ότι αυτό ε, πια επήγει όταν μιλάμε για δημοκρατικά καθιστώτα στην τρίτη χιλιετία και κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα. Μιλάω για το θέμα των αρμοδιοτήτων. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι αρμόδιος γιατί, πώς ε, λειτουργεί η επιτροπολογία, που σημαίνει τελικά ότι για την νομοθετική εξουσία, δηλαδή για εμάς τελικά, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε κάτι, ακόμα και για θέματα που είμαστε αρμόδιοι και όπου καλούμαθε τουλάχιστον να παρακολουθούμε τη δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας. Άρα δηλαδή το δεύτερο που θέλω να ζητήσω είναι λιγότερη περίπλοκο, περίπλοκη δομή. Λιγότερο περίπλοκη δομή. Και ε, να πω και κάτι για τους συναδέλφους μου εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε κάτι, ε, πραγματικά υποτιμούμε το πόσες αποφάσεις λαμβάνονται μέσω της επιτροπολογίας. Εγώ έχω κατά νου χιλιάδες ε, παραρτήματα τα οποία ε, συζητούνται στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, αλλά εκείνη η ουσία. Αυτή είναι η ουσία επί της καλούμεθα και εμείς να αποφασίσουμε. Άρα δηλαδή οφείλουμε ως ε, κοινοβούλιο να έχουμε καλύτερο έλεγχο και αναμφίβολα να μεριμνήσουμε, να συμμετέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αν τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι κατορθώσει να αλλάξει κάτι συγκεκριμένα έτσι ώστε ο απλός πολίτης, ο μέσος πολίτης να γνωρίζει περίπου το τι διαδραματίζεται. Αν το καταφέρει αυτό η Επιτροπή, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Ιρωνικά το λέω βέβαια αυτό, αλλά ξέρετε, το λέω ορμόμενοι από την εμπειρία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή βλέπω ότι δεν επιθυμεί κανείς άλλος ε, το λόγο, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για την τελική του τοποθέτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών για την τοποθέτησή τους που είναι ξεκάθαρη και εγώ επίσης περιμένω πώς και πώς να συνεργαστούμε και με τους σοσιαλδημοκράτες αλλά και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ναι, ακριβώς, όπως ελέγχθη. Είναι μεγάλο πειρασμό το να ξεκινήσουμε μια ευρύτατη συζήτηση για την επιτροπολογία και μελέτησα διάφορους κανονισμούς, εφαρμοστικές πράξεις, ε, κατεξοδότηση πράξεις και αναρωτιέται κανείς το κοινοβούλιο τι ρόλο έχει για την νομοθεσία. Τέλος πάντων, όχι, δεν θα ξεκινήσουμε τέτοια ευρύτατη κουβέντα. Αλλά αν συνεργαστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία και ευχαριστούμε και τη Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο, που σχολίασαν το θέμα των ε, εμπορικών μέτρων και θα μελετήσουμε τις ε, τροπολογίες όσο γίνεται καλύτερα και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται επίσης να ολοκληρώσει την εκτίμηση της καταστάσεως. Ευχαριστώ, οπότε και τώρα ολοκληρώνουμε για αυτό το σημείο, λέει ο Πρόεδρος, και όπως ε, είπαμε, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα. Τέλο πάντων τον Οκτώβριο πρόκειται να γνωμοτήσει η Επιτροπή. Και σα ευχαριστώ. Items uh, on the agenda, point number... Για να δούμε τώρα το επόμενο σημείο. Τα σημεία 6 και 7 αποτελούν μια κοινή συζήτηση όσον αφορά την ενισχυμένη εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατών μελών και από την άλλη μεριά τη δημοκρατία του Καζακστάν. Η σχετική συμφωνία υπεγράφει τον Δεκέμβριο του 2015 και προσωρινά τέτοιε σε εφαρμογή τον Μάιο πέρσι, το δε Νοέμβριο, ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο να συνενέσει, να εγκρίνει τέλο πάντων την ε, συνθήκη αυτή. Η ΑΦΕΤ ε, επίση εκλήθη να γνωμοδοτήσει και εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για τις δύο αυτές ε, εκθέσεις ο κύριος Μπορέλη είναι ο εισηγητής μας, ε, αλλά δεν μπόρεσε να προσέλθει στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα όμως βρίσκεται εδώ που θα σας πει τη γνώμη για τα δύο αυτά θέματα. Έχετε το λόγο κύριε Μπορέλη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τώρα αυτά τα σχέδια γνωμοδότηση όσον αφορά την ενισχυμένη εταιρική σχέση και τη σχετική συμφωνία αλλά και τη συνεργασία Ένωση και Καζακστάν. Για να θυμηθούμε τώρα το γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι σχέσεις των μερών. Η γεωγραφική θέση του Καζακστάν μετά την ανεξαρτησία έχουν καταστήσει τη χώρα αυτή ε, πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια της ε, πολιτικής μας για την Κεντρική Ασία. Και ε, επίσης αυτή η εταιρική σχέση ξεκίνησε το 1999. Έχουμε τώρα σημαντικές εξελίξεις της σχέσης μας γιατί το Καζακστάν θέλησε να ακολουθήσει μια διαδρομή προσέγγισης Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μια που ξέρουμε ότι χρειάζεται ευρύτερη συνεργασία. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα και η προηγούμενη φάση, το 2015 και από ό,τι είπαμε τώρα θα πρέπει να έχουμε αυτήν την ε, ε, προσωρινή ισχύ της συμφωνίας 15 με 17 όπως είπε ο Πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανανέωση της συμφωνίας. Είναι νέου τύπου συμφωνία για τις χώρες Κεντρικής Ασίας και μετά από αυτά τα ε, χρόνια συνεργασίας, τα 29 χρόνια, είπαμε ότι έχουμε αυτές τις ε, χώρες Κεντρικής Ασίας που τώρα θα ενταχθούν στην πολιτική γειτονία μας. Θα πρέπει έτσι επομένως να ρυθμιστούν οι σε σχέσεις με το Καζακστάν και τις ε, άλλες εκεί χώρες και έτσι να εξελιχθεί, να προχωρήσει η πολιτική γειτονία. Και θέλουμε η κυβέρνηση της ε, Αστάνα να σταθμίσει τις σχέσεις μαζί μας αλλά και τις σχέσεις με Κίνα και Ρωσία. Είναι μέλος της ε, Ευρασιατικής ε, Κοινότητας, έχει στρατηγική σημασία, είναι σημαντικός παίκτης στην Ασιατική Σκακέρα. Και θέλουμε επομένω να υπάρχει αξιοπιστία στην ανταπόκριση της ηγεσίας της χώρας και θα πρέπει να μάθουν τους μηχανισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό που μας βοηθά. Έχουμε επίσης πετρέλαιο και φυσικό αέριο το τρίτων των εξαγόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τους πουλάμε φαρμακευτικά, ε, μηχανήματα, πλαστικά, χημικά προϊόντα. 50% ε, επίσης των ξένων ε, επενδύσεων της χώρας είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην συμφωνία. Έχουμε 9 κεφάλαια, 87 άρθρα και μιλούμε για την ανταλλαγή των εμπορευμάτων, ε, ασχολούμεθα με, με τους τεχνικούς φραγμούς, τα φυτογειονομικά, στην σταθεροποίηση αυτών των ανταλλαγών, ε, κίνηση κεφαλαίων και άλλα θέματα ρυθμίζονται εκεί. Δεν αγνωστώ οικονομία της αγοράς, είναι η οικονομία σε μετασχηματισμό. Είχαμε τη συμφωνία του 2015, που πρόκειται να είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για τη χώρα. Θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητε ε, μεταρρυθμίσεις, ούτω ώστε να πλησιάσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη σχέσεις μας ότι αναπτύσσεται η οικονομία της χώρας, ε, και πλέον το πετρέλαιο και ε, το φυσικό αέριο δεν αρκούν για την ανάπτυξη της χώρας. Θα πρέπει επομένω να υπάρξει μετασχηματισμό της οικονομίας σε μια προτεραιότητα. Έχουμε αυτά τα 25 χρόνια της ανεξαρτησίας και αυτή την ευαίσθητη φάση της πολιτικής αλλαγής. Χρειάζεται να γίνει δημοκρατική αλλαγή και αυτό επίσης έχει σχέση και με τις διμερείς μας εμπορικές σχέσεις. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δύσκολο μέτωπο. Ε, έχουμε ξεκινήσει συγκεκριμένο διάλογο για αυτό, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τις συμφωνίες τελευταίας γενεάς. Και έχουμε τώρα τις ε, κινέζικες επενδύσεις που θα πρέπει να προσέξουμε να μην μας περιθωριοποιήσουν. Τώρα έχουμε ε, επίσης άλλα θέματα το σημείο Α αφορά τη σύνοψη της συμφωνίας, οπότε και αφορά τα οικονομικά και θέματα και αυτό αφορά το πώς θα αναδειχθεί ο soft η Ευρωπαϊκή στην Κεντρική Ασία, όπως ε, έχει ισχύσει και με άλλες συμφωνίες. Β. Έχουμε τη ε, μείωση των ε, διμερών ανταλλαγών, και οποίο αυτό αφορά το πόσο έχει καταρρεύσει η τιμή του πετρελαίου, με οι κυρώσει προς την ε, Ρωσία, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει βιωσιμή ανάπτυξη και καταπολέμηση της διαφθοράς σύμφωνα με τη στρατηγική μας ε, για την Κεντρική Ασία και ε, αυτό αφορά τα δεδομένα του 2016, το πρόβλημα που παραμένει εκρεμές γάμα προσεχώρησε η χώρα στον ΠΟΕ το 2015 και είχαμε εναρμόνιση της νομοθεσίας Έχουμε επίσης ε, ε, απομιμήσεις, πειρατεία ε, και διάφορες παραβιάσεις του δικαίου του copyright και είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρξει και εδώ ενισχυμένη συνεργασία. Δέλτα, όπως ήδη αναφέρθηκε, το η χώρα συμμετέχει στην Ευρασιατική Ένωση αλλά θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τους δασμούς τους όσον αφορά τις εισαγωγές Αλλιώς αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ τους εμπορευομένους. Επίσης έχουμε μία πλατφόρμα πληροφορική που αφορά τα κτηνιατρικά. Ε, επίσης ε, πρέπει να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι το να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους μέσω της συμφωνίας. ΣΥΓΜΑΤΑΦ έχουμε τώρα τις δημόσιες ε, συμβάσεις που θα πρέπει επίσης και αυτές να περάσουν από μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να προβλέπεται μια περίοδος ε, μεταβατική μιας πενταετίας τόσο ώστε να υπάρξει η σχετική απορρίθμιση. Ε, ζήτα τα... Ε, έχουμε κάποιες συλλήψεις συνδικαλιστών που δημιούργησαν αντιδράσεις από πλευρά Διεθνού Γραφείου Εργασία και μη κυβερνών οργανώσεων του Μάρτιο του 2016 και είχαμε και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου που λέει που ασχολείται ακριβώς με την ελευθερία της ε, έκφρασης. Ε, θεωρώ ότι πρόκειται να ε, έχουμε οικονομικό όφελος αυτή τη συμφωνία, αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια διαδρομή προσέγγισης της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών, υπάρχει κάποια πολυπλοκότητα θα πρέπει όμως να δούμε πώς με τέτοιου είδους διαδικασίες δεν θα υπονομεύεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Και σας ευχαριστώ συνάδελφοι για όσα είπατε. Και εμεί ε, ευχαριστούμε και πάω τώρα στις ε, πολιτικές ομάδες. Ε, πρώτα το ΕΛΚ, η κυρία Ρόβολ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπορέλη, να τον ευχαριστήσω για την ε, πολύ καλή δουλειά του. Ως ε, ΕΛΚ κατά περίπου 90% συμφωνούμε με την έκθεσή του. Το Καζακστάν είναι ένα σημαντικό εταίρο στην Κεντρική Ασία και το προσχέδιο του εισηγητή ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν ως ΕΛΚ θα συμφωνήσουμε με την επικύρωση της ε, Συμφωνίας Συνεργασίας. Και γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι οι διμερείς ε, σχέσεις ε, ε, θα πρέπει να ενισχυτούν, ε, να υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις συνεργασίας και εμείς πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει στο Καζακστάν βεβαίως να υπάρχουν και περισσότερες πολλές πολιτικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα τώρα να κάνω και μία άλλη παρατήρηση που αφορά στο σημείο G, δηλαδή το τελευταίο σημείο σε, αυτήν την, σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα σωστό να καλούμε μια ξένη χώρα Όχι, συγγνώμη, δεν αναφέρουμε στο Τζίλα το έκανα. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι δεν είναι σωστό να καλούμε μία χώρα να μην τηρεί τις υποχρώσεις της. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γνωρίζω ότι το Καζακστάν ε, συμμετέχει σε διάφορες συνεργασίες και νομίζω ότι είναι δύσκολο να τοποθετήσει κανείς σωστά όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας. Εμείς όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το Καζακστάν κάπως πρέπει να τα τακτοποιήσει όλα αυτά. Και η δεύτερη παρατήρησή μου, αυτή πραγματικά αφορά το σημείο υπαριθμών ε, G. Ε, όσον αφορά την ε, σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, εκεί θα ήθελα να έχουμε μια πιο θετική διατύπωση. Μπας περιπτώσει, θα καταθέσουμε τροπολογίες και κύριε Μπορέλη, αγαπητέ συνάδελφες, σας ευχαριστούμε πολύ καλή, για την καλή σας δουλειά, γιατί με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται κατά πολύ τη δουλειά των σκιωδών συντονιστών. Ο Ντέβιτ Μάρτιν, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, παρακαλώ. Η σκιώση ηγέτρια είναι η κυρία Μαρία Αρένα. Εγώ την αντικαθιστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπορέλη για τι εργασίε του πριν αρχίσω να διαβάζω τι δηλώσει τη Μαρία Μαρίας Αρένα. Αναγνωρίζουμε την στρατηγική σημασία του ρόλου του Καζακστάν. Είναι σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κεντρική Ασία και η διμερή συμφωνία, η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχιστεί. Όμω, η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι συνεκτική με τις ε, αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν εξακολουθεί να μας ανησυχεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφραση, ελευθερία ε, του συνεταιρίζεσθε, καθώ επίση και τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθούμε ε, στα ε, πρώτα συμπεράσματα του Δημερού διαλόγου ε, του περασμένου Ιουνίου που αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το θέμα. θα πρέπει η συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία, ε, να παρακολουθείται στενά σε συνδυασμό με, την, ε, με τις εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα και σύμφωνα με τους κανόνες του ILO, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για το ECR και τους φιλελεύθερους. Δεν βλέπω εκπροσώπηση. Η Γκουε. Παρακαλώ. Και ο Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ο σκιώδης ηγητής ε, δυστυχώς ε, σήμερα λείπει αλλά με παρακάλεσε να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις και ξέρετε έρχομαι από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όπου αυτή τη στιγμή συζητιέται η έκθεση όπου είμαι σκιώδης ηγητής ευθύς εξ αρχής θέλω να πω ότι πράγματι πρόκειται για ένα περίπλοκο και δύσκολο θέμα διότι δεν πρόκειται μόνο για τις εσωτερικές εξολήξεις στο Καζακστάν αλλά πρόκειται και για το πώς θα μπορέσουμε να προάγουμε την πολιτική και οικονομική συνεργασία με το Καζακστάν. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι οφείλουμε να δούμε πολύ προσεκτικά ποιες ακριβώς είναι οι διατάξεις ε, της ε, συμφωνίας. Μία συμφωνία που έχει τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή ήδη από το 2016. Δηλαδή, με τη διαδικασία επικύρωση απλά θέλουμε να καλύψουμε κάποιες υποχρεώσει μας και θέλουμε τώρα να δούμε ποιε είναι οι συνθήκε συνεργασία με το Καζακστάν και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Μάρτιν ότι στο Καζακστάν η κοινωνική κατάσταση, το θέμα των συνδικάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά ε, είναι θέματα που προκαλούν προβλήματα. Ένα θέμα που τέτοιε Επίση ε, είναι η σχέση όλων αυτών με το εμπόριο. Αυτό παίζει ρόλο με τις ε, χώρες του Ειρηνικού και της Ασίας. Άρα δηλαδή για να είμαστε πολιτικά συνεπείς ε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε και να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη, με τα Υπουργεία Εξωτερικών, αλλά και με τους εταίρους μας να καταλήξουμε σε μια συνεπή στάση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συνεπή συνέπεια στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί της ουσίας, για την έκθεση, θέλω να σας πω το εξής και ευχαριστώ τον κύριο Μπορέλη ε, που έθιξε το θέμα, ε, δηλαδή το ποια είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στη συνεργασία με την Ευρασιατική Ένωση. Ε, εδώ νομίζω πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να δώσουμε κάποια πιο οξία μορφή στην ε, γνωμοδότηση. Εμείς ευχαριστούμε να το κάνουμε. Και επίση, αυτά που σας είπα, το συσχετισμό με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους του Καζακστάν, αυτά πράγματι πρέπει να τα θέσουμε ως προϋπόθεση για την οικονομική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ε, η πράσινη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την πολύ, το πολύ καλό προσχέδιο γνωμοδότηση. Είναι πολύ καλό σημείο φετήριας. Δεν θέλω να επαναλαβώ όλα όσα υπόθηκαν μόλις τώρα. Να κάνω όμως μερικές παρατηρήσεις. Η... Και η δική μου ομάδα είναι διστακτική σε ό,τι αφορά την βελτίωση των ε, εμπορικών σχέσεων με το Καζακστάν, δεδομένου ότι τόσο το πολιτικό πανόραμα όσο και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν ε, δεν έχει βελτιωθεί, δεν έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα. Το Καζακστάν σίγουρα είναι μια χώρα η οποία έχει ε, καλύτερη απόδοση από άλλες ε, της ίδιας περιοχής και θα πρέπει να δούμε τη χώρα και στο γεωπολιτικό της περιβάλλον το έκανε ο εισηγητής σε σχέση με την Ουκρανία και την Ρωσία. Ε, είναι σε μια περιοχή που το Καζακστάν παίζει πολύ επικοδομητικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λυπούμαστε που η, συμφων... η ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία δεν περιλαμβάνει όρους ε, για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι έχει κάνει η χώρα αυτή ε, και να το συνδέσει με την εφαρμή της συμφωνίας. Ε, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τη μεταφορά τεχνολογίας και των πρώτων υλών, ε, έχουμε μια χώρα η οποία θα πρέπει επίσης να μας ε, διδάξει πράγματα γιατί ξέρει πάρα πολλά. Δεν πρέπει να είναι μονόδρομος η σχέση μας. Επίσης η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών ροών πρέπει να παρακολουθεί πολύ κοντά για να αποφύγουμε την ε, λεύκανση παράνομου χρήματος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Οπότε απευθύνομαι πλέον στην Κομισιόν. Ο Σουμέλης από ο κ. Σούμελης από την Γενική Ένση Trade θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον συγητή για το σχέδιο της έκθεσής του. Ε, όπως είχα την ευκαιρία να σας πω και όταν πρωτοσυζητήσαμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή, βεβαίω και το Καζακστάν είναι κατά πολύ ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Έχουμε έντονες εμπορικές σχέσεις με το Καζακστάν. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια μειώθηκε ε, όχι τόσο όγκος όσο η αξία των εμπορικών ανταλλαγών και αυτό οφείλεται στην τιμή του πετρελαίου. Πάντως τώρα έχουμε και πάλι, βιώνουμε ανωδική πορεία. Το Καζακστάν είναι βεβαίως ένα σημαντικός και αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος που έχουμε στην περιοχή και συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ε, γνωρίζετε, είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της προσχώρησης ε, του Καζακστάν στον ΠΟΕ και παράλληλα ε, συμφωνούμε και στηρίζουμε μια ενισχυμένη συμφωνία συνεργασίας με το Καζακστάν. Αυτή είναι η πρώτη ενισχυμένη συμφωνία συνεργασίας και εταιρική σχέσης ε, που ε, έχουμε διαπραγματευτεί με τις ε, πρώην χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες με άλλες χώρες στην περιοχή. Η συμφωνία στην οποία αναφέρομαι περιέχει πολλά και σημαντικά θέματα σε διάφορους τομείς και όλα αυτά συνδέονται και με το μηχανισμό ναι, αλλά ε, διευθέτησης, διευθέτησης διαφορών να συνεχίζω τώρα, τι να κάνω. Υπάρχει αυτός ο θόρυβος όπως ακούτε. I think it's uh, better to have uh, two minutes of break until we... Καλύτερα δύο λεπτά διάλειμμα μέχρι να δούμε τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται κάτι υπάρχει σήμερα. Το πρωί είχαμε πρόβλημα με τον κλιματισμό των διερμηνέων. Ε, στις καμπίνες των διερμηνέων. Τώρα όμως φαίνεται ότι λύθηκε το θέμα. Πρόκειψε άλλο. Δύο λεπτά διάρκεια. let's continue. So uh, let's hope that everything will be okay from now on. So Mr. Sobel is back to you and please uh, continue your thoughts. Yes, thank you very much. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν με τον μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης διαφορών για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα το οποίο υπάρχει στο Καζακστάν και ίσως και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε και στο να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στο Καζακστάν, να υπάρξει ε, μεγαλύτερη και καλύτερη διαφεροποίηση στην παραγωγή της χώρας. Έγινε λόγος γι' αυτό σήμερα. Έγινε λόγος για τα ενεργειακά προϊόντα. Και τώρα ίσως θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια και για το τι προτείνει το σχέδιο της έκθεσης. Στο σημείο Β. Εκεί υπάρχει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ενισχύσουν, να στηρίξουν τις αρχές του Καζακστάν ε, για να ε, στηρίξει, να εφαρμόσει και αυτή τις αρχές της διαφάνειας. Εμείς έχουμε κάποια σχέδια που αφορούν στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τον Νοέμβρη προβλέπεται ότι στο Καζακστάν θα μεταβούν εμπειρογνώμονες για να δώσουν και πρακτική εμπειρία και πρακτικές συμβουλές στους αρμόδιους υπαλλήλους στο Καζακστάν. Υπάρχει και η ανάλυση χάσματος, αυτή ολοκληρώθηκε τελικά και αυτή αποτελείται από διάφορες τομείς της συμφωνίας, ε, δηλαδή ε, προτιθέμεθα να εξετάσουμε ε, ποια είναι η νομοθεσία που ισχύει στο Καζακστάν και τι είδου αλλαγέ ε, πρέπει να λάβουν χώρα έτσι ώστε το Καζακστάν να μπορεί να εκπληρεί τι διάφορε υποχρεώσει που προβλέπονται στη συμφωνία. Αυτέ είναι δύο προπαρασκευαστικέ πράξει ε, που έχουμε κατά νου για να μπορεί και το Καζακστάν να εφαρμόζει καλύτερα τι υποχρεώσει του. Πάμε στο σημείο υπερθμών C. Εκεί γίνεται λόγο κυρίω για τα πνευματικά δικαιώματα δικαιώματα, σχετικές υποχρεώσεις και υπάρχει μία αναφορά ε, στο καθεστώς που ισχύει στη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς το έχουμε δείξει στις αρχές του Καζακστάν και αυτές μας διαβεβαίωσαν ότι θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 της ενισχυμένης συμφωνίας συνεργασίας και εταιρικής σχέσης και γίνεται και μια συζήτηση στους αρμόδιους φορείς της Ευρασιατικής Ένωσης, ίσως για να ε, τροποποιηθεί Ε, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου τις υποχρώσεις του Καζακστάν και να είμαστε και σίγουροι ότι θα τηρούνται αυτές οι υποχρώσεις. Όσον αφορά στο σημείο υπερθμών E, ε, εδώ πρόκειται για θέματα εμπορικά. Τα συζητήσαμε αυτά με τις αρχές του Καζακστάν το Μάρτιο, όταν είχαμε την πρώτη επιτροπή που ασχολήθηκε με εμπορικά θέματα. Είναι σημαντικό για, τους, ε, για το Καζακστάν να συμμετέχει στο σύστημα Traces. Ε, βεβαίως με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εφαρμογή των, ε, της συμφωνίας SPS και αυτό που έχει σημασία για μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το Καζακστάν ε, θα δέχεται τα διμερεί επιστοποιητικά SPS την, τα επιστοποιητικά που αφορούν στη λήξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τώρα την ε, Ευρασιατική Ένωση, έχουμε την εξή κατάσταση. Το Καζακστάν έχει προσχωρήσει στον ΠΟΕ με ένα συγκεκριμένο σχέδιο ε, δασμών και προτάσεις για δασμολογικές κατηγορίες. Βεβαίως και υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις και όροι, αυτή είναι πολύ πιο ευνοϊκή για το Καζακστάν από ό,τι ισχύουν γενικότερα για την Ευρασιατική Ένωση. Το Καζακστάν στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη των ΠΟΕ είπε ότι στο μέλλον επιθυμεί να προβεί σε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε αυτά τα οποία εφαρμόζει να είναι συμβατά με το ενωσιακό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ισχύουν δασμοί στο Καζακστάν, αυτοί ε, τους οποίους έχουμε διαπραγματευτεί. Και στο μέλλον ε, θέλει το Καζακστάν να εκμεταλλευτεί αυτά που προσφέρει ο ΠΟΕ, ε, να αλλάξουν οι υποχρεώσεις τους. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ε, θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφερθεί απαραίτητη αποζημίωση, αν κριθεί κάτι τέτοιο απαραίτητο. Και τέλος, όσον αφορά το σημείο υπαρθμών G, που έχει σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα και το σεμβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ Έχουμε εσωτερική συνεργασία και με άλλους συναδέλφους, κυρίως από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, αλλά και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και αυτό το κάνουμε για να ενισχύσουμε τη μόχλευση που υπάρχει για το Καζακστάν και να διασφαλίσουμε ότι το Καζακστάν θα τηρεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Ήδη έχουμε ε, αφιερώσει πολύ χρόνο. Είχαμε την πρώτη Επιτροπή Εμπορίου και Συνεργασίας, ε, η οποία συνεδρίασε παράλληλα το Μάρτιο ε, και εκεί τέθησαν διάφορα θέματα έναντι των αρχών του Καζακστάν. Και με αυτή την ευκαιρία οι αρχές του Καζακστάν μας ενημέρωσαν ότι επιθυμούν να αναθεωρήσουν και πάλι το νόμο περί συνδικάτων έτσι ώστε ο νέος νόμος να συμβαδίζει να είναι σε αρμονία με τις διατάξεις του ILO και τις διεθνείς προδιαγραφές, τους διεθνείς κανόνες. Ε, προτιθέμεθα λοιπόν αυτό το θέμα να το παρακολουθήσουμε πολύ πιο προσεκτικά στο μέλλον και αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ κατά τους επόμενους μήνες στις διμερείς επαφές που θα έχουμε με το Καζακστάν. Αυτά τα σχόλια είχα να κάνω κύριε Πρόεδρε όσον αφορά στο σχέδιο της εκτής του κυρίου Μπορέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Επιστρέφουμε στον εισηγητή για να κλείσουμε έτσι τη συζήτηση. Τη συζήτηση Πρώτα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τα όσα ανέφεραν. Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζετε, όσον αφορά μια έκθεση, έχουμε ε, περιορισμό. Δεν μπορούμε να γράψουμε όσα ε, θα μπορούσαμε να γράψουμε. Γνωρίζουμε τι ισχύει για το Καζακστάν. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο χώρο, να πούμε πολύ περισσότερα. Όμως ε, ε, πρέπει να κάνουμε μία σύνθεση των απόψεων και ε, θα πρέπει περιληπτικά να φέρουμε όλα όσα εθίγησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την σημασία της συνεργασίας μας με την χώρα μέσα στο γεωπολιτικό περιβάλλον της χώρας. Με τις τροπολογίες ε, βεβαίως το κείμενο πρόκειται να έρθει πιο κοντά και να συγκεραστούν οι απόψεις των ε, συναδέλφων. Και ακριβώς ε, το τελευταίο σημείο που αναφέρθηκε είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ενεργοποίηση αυτής της προσωρινής συμφωνίας σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Οπότε βεβαίως και συμφωνώ επ' αυτού με τους συναδέλφους. Και τους ευχαριστώ και πάλι. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά και ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που συμμετέχουν στη συζήτηση. Έχουμε Τετάρτη Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα καταληκτική ημερομηνία για τις ε, προθεσμίες 25 του μηνός πρόκειται να συζητήσουμε, να ψηφίσουμε το σχετικό ψήφισμα σχετική έκθεση. Αυτά για το σημείο τούτο, το 6 και το 7. Και τώρα πάμε στο 9 που είναι η ανταλλαγή απόψεων ε, με την Επιτροπή να εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, τι γίνεται με αυτό το εργαλείο τη μακροοικονομικής συνδρομής. Και έχουμε την έκθεση της Επιτροπής προς Συμβούλιο και Κοινοβούλιο που αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση αυτής της ε, σύνδρομης του, την έκθεση του 2016. Εκεί ε, αναπτύσσονται τα της ε, υλοποίησης ε, αυτών των προγραμμάτων σε Γεωργία, Ιορδανία, Κυργισία, Μολδαβία, Δινησία και Ουκρανία. Και τώρα, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Οντρία έχουμε τον κύριο Λέναρτ, ο οποίο είναι ο τμήματάρχης για την μακροοικονομική βοήθεια της ε, Γενικής Διεύθυνσης για Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και μας παρουσιάσει τα της εκθέσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και αναφέρατε θα σας ε, παρουσιάσω σύντομα το τοπίο που αφορά την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για τις 3 του 2016. Να δούμε δηλαδή πώς ε, σήμερα έχουμε τον πράγμα, πώς έχει υλοποιηθεί αυτή η συνδρομή. Το 2016 χαρακτηρίζεται από συνεχή πρόοδο όσον αφορά ε, τα σχετικά προγράμματα για τις χώρες που αναφέρατε, Γεωργία και για την Ισία και Ουκρανία. Βέβαια, κάποιες εκταμιεύσεις έπρεπε να καθυστερήσουν για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της ε, Ένωσης πίεσης. Η συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική δυσκολία για κάποιες γειτονικές χώρες ε, μας οδήγησε σε έγκριση δύο πράξεων σε την Ισία και η Ορδανία. Επίσης είχαμε μια νέα πράξη που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Μολδαβία. Και τώρα, να σας περιγράψω το τοπίο του πώς έχει σήμερα ε, η κατάσταση ανά χώρα. Το 2016 είχαμε την τελευταία δόση αυτή της βοηθείας που αφορά την εκεργησία. Τότε είναι επόμενος η σχετική εκταμίευση και τότε ολοκληρώσαμε αυτήν την ε, πράξη που ήταν εξαιρετικό χαρακτήρα γιατί είπαμε ότι η Κυριασία είναι εκτός του συνήθους α, πεδίο εφαρμογή αυτού του εργαλείου. Αλλά είπαμε ότι θα πρέπει να προβούμε σε αυτή την πράξη για να βοηθήσουμε την, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Και ε, επίσης είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά τα σχετικά με την αιρεσιμότητα ε, της τελευταίας δόσης του 16 φέτος. Επίσης, ολοκληρώσαμε την τελευταία πράξη που αφορά την ε, γεωργία. Η τελευταία δόση του 13 εκταμιεύθηκε τον Μάιο. Όμως, το το τοπίο είναι δυσχερές και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ε, ενέκρινε ένα τρίτες πρόγραμμα ακόμα είναι πάρα πολύ ευάλωτη η χώρα όσον αφορά ε, την, το ίσως γεωπληρωμών και ζητήθηκε μια ανανέωση αυτής της ε, συνδρομής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει την έγκριση αυτής της πράξης Ήδη συζητήσαμε με την Χρηματοοικονομική Επιτροπή. Υπάρχει ε, σύμφωνη γνώμη για να υπάρξουν ε, και άλλες τέτοιες πράξεις ενίσχυσης προ την υγειοργία και θα δείτε τι προτάσεις μας αρχάς του Οκτωβρίου προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επίσης ε, θα έχουμε μια πράξη που θα φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ μάξιμου στα πλαίσια τη αρχική βοήθεια των 10 εκατομμύρια. Για τη Γεωργία τώρα, στη συνέχεια της κρίσης της ε, Συρίας, είχαμε επιβράδυνση τη ανάπτυξη. Ε, άλλο 2% το 2016 και αυτό ήταν ε, ο πιο αργός ανάπτυξη ανάπτυξης το 2010 για την χώρα. Επίσης, σήμερα υπάρχει έλλειμμα στις τρέχουσες μιλούμε για 9% και φτάσαμε στο 13% δηλαδή του ΑΕΠ. Σε αυτά τα πλαίσια η Επιτροπή πρότεινε μια δεύτερη πράξη συνδρομής για την ε, Γεωργία 200 εκατομμύρια ως δάνεια. Αυτό εγκρίθηκε από τους συνομοθέτες τον Δεκέμβριο του 2016. Οι δε διαπραγματεύσεις όσον αφορά το σχετικό μνημόνιο μόλις ολοκληρώθηκαν και αυτό το μνημόνιο πρόκειται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα. Οπότε και έτσι θα μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε την πρώτη δόση ε, τέλη του Οκτωβρίου. Έχουμε την κοινή δήλωση Κοινοβουλή Συμβουλική Επιτροπή στα πλαίσια αυτής της ε, πράξης. Οπότε και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει κάποιο είδους ε, συνέχεια και η Επιτροπή πρόκειται να παρακολουθεί την εξέλιξη όταν η πράξη που αναφέραμε, η τωρινή δηλαδή, πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, για την Τινησία. Για την Τινησία ε, ε, είναι συγκρατημένος ο ρυθμός ανάπτυξης, ευάλωτη είναι το ισοζύγιο πληρωμών, 9% το έλλειμμα περίπου και όταν ολοκληρωθεί η πρώτη εξολόγηση του προγράμματος του ΔΕΛΤΑ πρόκειται να κάνουμε την αποτίμηση του πρώτου προγράμματος οπότε και θα εκταμιεύσουμε την ε, τελευταία δόση των 100 εκατομμυρίων προς την χώρα στα τέλη Ιουλίου. Η δεύτερη πράξη για το σύνολο των 500 εκατομμυρίων θα καλύπτεται από τρεις πράξεις 200, 150 150 και αυτό θα γίνει κατόπιν της υπογραφής του Μνημονίου τον Απρίλιο. Και πρόκειται έτσι να έχουμε και την εκκύρωση των σχετικών ε, εγγράφων και συμφωνίων τον Ιούλιο. Η εκταμείευση τις πρώτες ε, δόσεις, δεν ε, εξαρτάται από κάποιους ε, όρους, κάποια ρεσιμότητα και θα γίνει επομένως η εκταμείευση τον Σεπτέμβριο. Ουκρανία. Η μακρογνωμική σταθεροποίηση προχωρεί. Όμως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για την οικονομία της χώρας, γιατί είναι πάρα πολύ μετάβολη η κατάσταση και έχουμε το 2019 προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές. Οπότε υπάρχουν διάφοροι ε, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και επίσης η χώρα έχει προβλήματα εξωτερικές πληρωμές μέσω πρόθεσμα. Και ε, κατόπιν της κρίσης του 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ενέκρινε μια συνδρομή 3,4 δισεκατομμύριων. Σύνολο 2,8 δις ήδη έχουν εκταμιευθεί και στις 16 Μαρτίου μετά κάποιες καθυστερήσεις που αφορούν την υλοποίηση των προϋποθέσεων για τις μεταρρυθμίσεις μπορέσαμε να εκταμιεύσουμε τη δεύτερη δόση των 600 εκατομμυρίων στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος της συνδρομής. Έχουμε επίσης την τρίτη ε, δόση εάν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται εγκαίρως. Θα συνεχίσει το πρόγραμμα του Δελτανιτάς και θα πρέπει να δούμε το ότι ήδη πληρούνται τα δύο τρία των προϋποθέσεων και στις επαφές μας με την χώρα τονίσαμε το πόσο σημαντικό είναι να επιταχυνθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Αλλιώς ε, δεν θα γίνει εκταμείευση της τρίτης πράξης. έχουμε αυτό, αυτή την περίοδο των 2,5 ετών που εκπνέει τον Ιανουάριο του 18. Τέλος, Μολδαβία. Εδώ υπάρχουν δυσκολίες τα τελευταία δύο χρόνια και οικονομικά και πολιτικά. Γιατί είχαμε ένα μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο σχετικά με απάτες, το οποίο ξέσπασε τον 2014. Οπότε και έτσι επιβραδύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα γιατί είχε προβλήματα δημοσιονομικά και ζήτησε και έλαβε υποστήριξη η χώρα από το ΔΝΤ Ξεκίνησε επομένως ένα τριετές πρόγραμμα του ΔΝΤ. Επίσης ζητήθηκε και μακροοικονομική συνδρομή από εμάς. Και τον Ιανουάριο του 2017 κάναμε τη σχετική πρόταση για μια πράξη 100 εκατομμυρίων, 60 εκατομμύρια δάνεια και 40 εκατομμύρια επιχορηγήσεων. Αυτή η συνδρομή πρόκειται να εκταμιευθεί σε τρεις δόσεις. Έχουμε κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις για κάθε δόση. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να ισχυροποιηθεί η κυβέρνηση, να καταπολεμηθεί η διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, μεταρρυθμίσεις και στα ενεργειακά, επίσης και στα πλαίσια της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και οι εμπορικές συμφωνίες να υλοποιηθούν και είχαμε τροποποίησει τις σχετική μας απόφασεις για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά το σχετικό μνημόνιο. Να γίνουν μεταρρυθμίσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να κατοχυρωθεί ο πλουραλισμός στα ΜΜΕ. Επίσης, είχαμε μια κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων σε σχέση με το ότι θα πρέπει να εκδημοκρατιστεί η χώρα, να υπάρχει πολυκομματισμός και κρατός δικαίου. Αυτά όλα είναι προϋπόθεση για να χορηγηθεί αυτή η οικονομική βοήθεια. Και σύμφωνα με αυτές τις δηλώσεις και διάφορες ε, πρωτοβουλίες, αλλαγή του εκλογικού νόμου κλπ. Παρακολουθούμε το πώς θα πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις εμείς και οι υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Δεν θα πρέπει οι αρχέ της χώρας να τηρήσουν τα όσα έχουν δεσμευτεί προς τους διεθνεί ε, εταίρου τη της χώρας και προ εμά. Οπότε θα σα ενημερώσουμε για το τι γίνεται για κάθε δόση, για κάθε εκταμίευση, για αυτή την ε, οικονομική συνδρομή. Όπω γνωρίζετε, το χρονικό πλαίσιο προβλέπει η σχετική απόφαση να υπογραφεί από τους Πρόεδρους Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στην Σύνοδο του Σεπτεμβρίου και κατόπιν αυτής της επίσημης ε, έγκρισης της σχετικής απόφασης η Επιτροπή θα έχει εξουδοτηθεί για να ολοκληρώσει το μνημόνιο. Έχουν ήδη αρχίσει για το μνημόνιο διαπραγματεύσει με τη χώρα. θα πρέπει βέβαια να προηγηθεί η κύρωση από κοινοβουλίου και μετά να ισχύσει, να τεθεί σε φορμή άλλο το μνημόνιο. Ε, πρόκειται να σας ενημερώσουμε για το σχετικό σχέδιο του κειμένου και θα γίνει διαβούλευση με κοινοβούλιο και συμβούλιο. Θα σας στείλουμε το σχετικό σχέδιο κειμένου πριν αυτό εγκριθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εδώ θα βάλω τελεία. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, παρουσίαση. Ε, καταρχήν θα δώσω το λόγο στους ε, μόνιμους εισηγητές των χωρών, των δικαιούχων χωρών. Δεν είναι όλοι εδώ. Αλλά πολλοί αντικαθίστανται. Ε, για τη Γεωργία Κυριατάκουλα, για την Ιορδανία ο κ. Μορέλ, για την Κυρική, Δημοκρατία, κυρία Έλλη, και για την Μολδαβία η Σολίν Μόισα. Η κυρία Λαλόντ για την Τινησία είναι παρούσα. Δεν μπορεί να θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να θέσω μερικές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για την Ισία. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποιες ε, ε, εκταμιεύσεις έχουν γίνει στο πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα και επίσης τι γίνεται με τις επαφές με τις ε, ε, ε, αρχές της Τινησίας. Δεύτερον, παρατηρητές ανησυχούν για την οικονομική κατάσταση της Τινησίας. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πολιτική αστάθεια. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Έχετε διαπιστώσει βελτιώσεις στην εκταμίευση των διαφορετικών δόσεων της ενίσχυσης, της συνδρομής. Ευχαριστώ. Uh, very... Απάντηση. Ε, συγγνώμη, ο πρόεδρος. Ο κ. Βαλέσα είναι ο εισηγητής για την Ουκρανία, επίσης ε, δεν είναι εδώ. Ε, περνάω στους συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων για, την, για το ΕΛΚ, η Γκοντελίβ. Συντονίστρια του ΕΛΚ. Ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν πρόσεχα. Περνάω στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Αλέσια Μόσκα. Παρακολουθήσαμε τι εξελίξει στι διάφορε χώρε και βεβαίω και εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω περισσότερα πράγματα για την Τινησία. Γιατί η Τινησία είναι μια χώρα η οποία μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αυτό ε, διότι γίνεται πολλή δουλειά από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί το θέμα του, το πρόβλημα του μεταναστευτικό. Ευχαριστώ. Το ECR δεν εκπροσωπείται. Η φιλελεύθερη. Ε, εντάξει. Γκουέ, ο κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Κομισιόν για τι πληροφορίε που μα έδωσε Ε, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, θα ήθελα πιο λεπτομερή πληροφόρηση για την ε, τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν λάβει αυτές οι χώρες, που έχουν αναλάβει αυτές οι χώρες. Κάθε φορά που συζητούμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέμε ότι θέλουμε να έχουμε σαφή εικόνα για το κατά πόσον η μικροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έχει συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης στις χώρες αυτές. Θα μπορούσατε τακτικά, ενδεχομένως γραπτός, να μας ενημερώνετε για το ποια πρόοδος έχει γίνει. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε στην τρίτη δόση στην Ουκρανία. Είπατε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά τι προβλήματα τι ακριβώς δεν έχει τηρηθεί, τι ακριβώς δεν έχει υλοποιηθεί. Γιατί ε, θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά τα ζητήματα στο μέλλον. Και εγώ επίσης θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για την Τινησία και για τη Μολδαβία. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση στην Μολδαβία δεν έχει αλλάξει και πολύ, παρόλο που το, η, η συνδρομή ε, φτάνει. Χρειαζόμαστε επίσης να κάνουμε μια πολύ βαθιά συζήτηση για το μνημόνιο. Πριν η υπογραφή στην Σύνοδο της Ολομέλειας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι συντονιστές. Και κ. Σούστερ έχει στήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Σόλτς. Συγκεκριμένα για την Ουκρανία. Θέλω περισσότερες πληροφορίες. Ε, η εκταμείευση της ε, μακροοικονομικής συνδρομής συνδέεται με συγκεκριμένους όρους. Τώρα, κατά πόσον αυτοί εκπληρούνται στην Ουκρανία, εγώ έχω πολλές αμφιβολίες. Εξακολουθεί να υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, ε, καμία δίωξη. Οι ολιγάρχες εξακολουθούν να ασκούν μεγάλη επιρροή στο κόμμα και αυτό ε, έχει ως αποτέλεσμα ότι στο κοινοβούλιο ε, νομοσχέδια τα οποία περικόπτουν τα συμφέροντα των ολιγαρχών απλά απορρίπτονται. Πιστεύαμε ότι θα υπάρξει βελτίωση στην οικονομία, αλλά μεταξύ η, η, η μαύρη αγορά, η μαύρη οικονομία έχει επεκταθεί και αυτή πάρα πολύ και μόνο αυτό, αλλά προστίθεται και μαζική ε, διαφυγή κεφαλαίων από την Ουκρανία που καταλήγουν στην Κύπρο και σε άλλες χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ και εγώ, τι έγινε τελικά με τους όρους, πληρούνται αυτοί ή όχι και τι θα γίνει με την τρίτη δόση. Εσείς υπενηχθήκατε ότι θα μπορούσε να μην λάβει χώρα η τρίτη δόση, η εκταμείευση της. Ε, εγώ πιστεύω ότι δεν εκπληρούνται οι όροι. Εσείς πώς καταλήγετε ότι οι όροι πληρούνται και ότι θα μπορούσε πράγματι να εκταμιευτεί η Ευχαριστώ. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Πριν τον δώσω στην Κομισιόν, θέλω να κάνω κι εγώ ένα προσωπικό σχόλιο και δύο ερωτήσεις. Το σχόλιο αφορά την συμφωνία με την Μολδαβία. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις πληροφορίες που μας δώσατε. Το σχόλιο μου λοιπόν είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τηρήσετε αυτή τη θέση της Κομισιόν την οποία μας διαβάσατε. Γιατί αυτή η θέση έχει ήδη συζητηθεί και εδώ στο Κοινοβούλιο Μακρόν Δυστυχώς δεν ακούμε πολλά καλά νέα από το Κισινιόφ. Μόνο ανησυχητικές ειδήσει ακούμε από τη Μολδαβία. Οπότε θα πρέπει να παραμείνουμε ε, σταθεροί στην θέση την οποία μας διαβάσατε και την οποία έχουμε συζητήσει. Και δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Η βελτίωση ε, της ε, ενημέρωσης από την DG ECFIN ε, εκ μέρους της ε, ε, του Κοινοβουλίου ε, και την ε, μεταβίβαση όλων των εγγράφων που δεν έχουν σχέση με την επιτροπολογία για αυτό το θέμα. Ο κ. Λάγκε είχε στείλει μια επιστολή στις 12 Ιουλίου στον Επιτροπό κ. Μοσκοβισή για το θέμα της ενημέρωσης για τα σημειώματα και τα ανεπίσημα έγγραφα. Ο... Αυτό αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να στέλνονται όχι μόνο στο όργανο το οποίο τα ζητά, αλλά και σε όλους τους συνομοθέτες. Δεύτερη ερώτησή μου. Ε, στην έκθεση του 2016 αναφέρονται ενδεχόμενα προγράμματα για το 2017 για ένα αριθμό χωρών. Αρμενία, Γεωργία και Αίγυπτο βασικά και ενδεχομένως ε, επακόλουθες πράξεις για την, πράξη για την Ιορδανία. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται η κατάσταση για αυτές τις τέσσερις χώρες. Αυτά. Έχετε το λόγο κύριε Λέναρτς. Ε, thank you, Mr. Θα δώσω... Θα ξεκινήσω από την Τινησία. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις καθυστερήσεις. Πράγματι, παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην εκταμίευση της συνδρομής προς την Τινησία. Πρώτον, άργησαν οι Τινήσοι να επικυρώσουν τα έγγραφα. Εν τω μεταξύ έλαβαν χώρα και εκλογέ, πέρσι νομίζω και αυτό καθυστέρησε έτσι περαιτέρω την χωρίση της συνδρομής. Τέλος, ορισμένα από τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που συνδέονταν με τις δόσεις έπρεπε πρώτα να εφαρμοστούν προκειμένου να γίνει εκταμίευση. Τελικά, σε συμφωνία με την Επιτροπή των Κρατών Μελών που ασχολείται με το θέμα, αποθεσμεύθηκε η τελευταία δόση της ε, πρώτης ε, του ε, ε, πρώτου τμήματος 100 εκατομμύρια υπό έναν όρο και η εκταμίση αυτή είναι τον Ιούλιο. Ο συνάδελφός μου μάλιστα μου λέει ότι ε, έχει σταλεί και ενημερωτικό σημείωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα και στο Συμβούλιο βέβαια. για την, για την τρέχουσα, ε, για το τρέχον τμήμα της ε, συνδρομής όμως. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί από ό,τι φαίνεται, έχει γίνει επικύρωση. Ε, η πρώτη δόση έχει ως όρο μόνο την συμφωνία με το Διεθνές Ταμείο, οπότε σύντομα θα αποδεσμευθεί υπό την προϋπόθεση ότι ε, οι όροι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα, θα πληρούνται. Ε, εμείς δεν έχουμε δικούς μας όρους δηλαδή α, και δεν έχουμε και κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα πληρωθούν αυτοί οι όροι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η δεύτερη δόση θα αποδεσμευθεί μέχρι το τέλος του 2017. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, όπως σας ανέφερα, παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις ε, με την δεύτερη δόση του τρίτου τμήματος 600 ε, εκατομμυρίων. Τελικά η Κομισιόν ε, έκρινε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και προέβη στην εκταμίευση νομίζω το Μάιο Η τρίτη δόση, όπως ανέφερα, είναι πιο περίπλοκο ζήτημα. Ε, στις 4 Ιανουαρίου 2018 λίγη αυτή η ε, πρωτοβουλία, λίγη η, ζωή αυτού του τμήματος συνδρομής. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι των υποχρεώσεων έχει υλοποιηθεί, αλλά ε, υπάρχουν και μέτρα που δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουμε μέτρα ε, για, την, για το πόθεν έσχεση των δημοσίων λειτουργών, μια επιγραμμική βάση δεδομένων για, την, για τα ονόματα των ιδιοκτητών εταιριών των πραγματικών δικαιούχων, ε, θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς ε, ε, και ανάκτησης ποσών. Ε, Επίση υπάρχει μια κρεμότητα σε ό,τι αφορά την πρώτη αξιολόγηση ε, και επιπλέον κάποια μέτρα στρέβλωση του εμπορίου τα οποία θα πρέπει να ανακληθούν ε, και μπορεί αυτό να δημιουργήσει θέματα. Επιπλέον στο χρηματοοικονομικό τομέα έχουμε την θέσπιση ενός κεντρικού μητρώου πιστωτών η οποία πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί μάλλον. Αυτά είναι οι λεπτομέρειε ό,τι αφορά ε, τα, τις ε, μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν από την Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά την Μολδαβία, επιβεβαιώνω μόνο αυτό που είπα προηγουμένω. Κατόπιν της επίσημης υιοθέτηση ε, μέσα σε Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις αρχές Μολδαβίας για το μνημόνιο, ε, ως τμήμα της διαδικασίας θα γίνει η αξιολόγηση των πολιτικών προϋποθέσεων, τις οποίες ανέφερα και προηγουμένως. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία μεταξύ Κομισιών και, Επιτροπή, και Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και προφανώς ε, ε, το αποτέλεσμα θα επηρεάσει την απόφαση του κατά πόσο θα προχωρήσουμε με το μνημόνιο. σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση εγγράφων. Την... Ε, θα ήθελα να ε, επιβεβαιώσω ότι λάβαμε την επιστολή του Πρόεδρου της Επιτροπής του κ. Λάγκε. Ετοιμάζουμε την απάντησή μας αυτή τη στιγμή. Χαιρόμαστε που ο πρόεδρος επιβεβαιώνει την, ε, επιτρο... την συμφωνία μεταξύ της ΕΙΝΤΑ και της ε, Κομισιόν, ε, της ΕΚΦΙΝ συγκεκριμένα. Θα συνεχίσουμε να σας διαβιβάζουμε όλα τα έγγραφα τα οποία έχουμε συμφωνήσει στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε την λειτουργία του Register for Committee Proceedings, του, του, του εργαλείου, του ηλεκτρονικού εργαλείου, που είναι ένα ηλεκτρονικό μητρό, μέσω του οποίου η Επιτροπή ΙΝΤΑ ε, ενημερώνεται για τα έγγραφα τα σχετικά με το μνημόνιο, με τα μνημόνια. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι τα, σε τα ανεπίσημα έγγραφα, η Κομισιόν θα πρέπει να τα στέλνει μόνο στο όργανο το οποίο τα ζητά. Αν δηλαδή τα ζητά το, κοινο, το Συμβούλιο, θα πρέπει τα non-papers αυτά να στέλνονται μόνο στο Συμβούλιο, αν τα ζητά το Κοινοβούλιο να στέλνονται μόνο στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό συνάδει με την ίση μεταχείριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ε, την ε, πληροφόρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικέ δράσεις για φέτος, ήδη σας είπα ότι θα γίνει μια επακόλουθη πράξη ε, για την γεωργία. Είμαστε, έχουμε προχωρήσει αρκετά στην προετοιμασία των νομικών εγγράφων. Θα τα λάβετε ενδεχομένως στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτή η πράξη για τη Γεωργία θα είναι παρόμοια με την προηγούμενη 45 εκατομμύριων ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες που αναφέρατε, η Ορδανία, σύμφωνα και με την δήλωση, κοινή δήλωση Κομισιών Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης πράξης, ε, θα εξεταστεί η δυνατότητα μια επακόλφης πράξης, τρίτης συγκεκριμένα, αλλά αυτό μόνο όταν λήξει, μάλλον όταν υλοποιηθεί η δεύτερη. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει εκταμιεύσεις για την τρέχουσα πράξη. Σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες τώρα, Αρμενία και Αίγυπτος. Ε, αυτά είναι ακόμα υποθέσεις. Ε, η Αρμενία δεν έχει υποβάλει έτοιμα ακόμα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα λάβουμε εμείς κάποια πρωτοβουλία. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την Αίγυπτο. Δεν έχει προκύψει κάποιο αίτημα εκ μέρους της Αιγύπτου για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Ήδη βρίσκονται σε πρόγραμμα του Δουνουτού, μεγάλου ύψους, χρηματοδοτούνται πλήρως από εκεί και δεν χρειάζονται περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Και εμεί σα ευχαριστούμε. Έχουμε και δύο ερωτήσεις από ε, αυτών που ελέγχθησαν. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Έχουμε εξάλλου και χρόνο. Ε, δίνω πρώτο λόγο στον κύριο Σόλτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση σχετικά με την Ουκρανία μετά από αυτά που είπατε. Μας είπατε ότι το χρονικό πλαίσιο είναι αρκετά περιορισμένο, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2018 τελειώνει η τρίτη δόση. Ποιο είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα ελέγξετε κατά πόσον πληρούνται οι όροι όχι. Πότε θα πάει επί τόπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι θα πρέπει να τοποθετηθούμε εμεί και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Θα πρέπει να ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε ε, τι γίνεται τελικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Και άλλη μια ερώτηση από τον κύριο Σούστερ. Ε, κοιτάξτε, είναι περισσότερο παρατήρηση αυτή που θέλω να κάνω. Το ερώτημα που σας έκανα δεν το απαντήσατε. Εγώ δεν ήθελα να μου απαριθμίσετε τους όρους, αλλά ήθελα να μάθω τι ήταν εκείνο που παρακίνησε την Επιτροπή και την οδήγησε στο να καταλήξει ότι τώρα πληρούνται ή δεν πληρούνται οι όροι. Τώρα, τα άλλα, τους όρους, τα διαβάζω και μόνη μου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ε, για την Ουκρανία, εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Οι δομές των ολιγαρχών άλλαξαν, ναι ή όχι και η καταπολέμηση της διαφθοράς προχώρησε, ναι ή όχι. Για μένα αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα και δυστυχώς δεν τοποθετηθήκατε ικανοποιητικά επ' αυτού. Και εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον πριν εκταμιευτεί η τρίτη δόση, το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί σωστά και όχι έτσι να μας λέτε γενικόλογα ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι όλοι πληρούνται ή δεν πληρούνται, αλλά να μας εξηγείτε και να τεκμηριώνετε την άποψη σας. Αυτό με ενδιαφέρει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις δύο ερωτήσεις και για άλλη μια φορά λοιπόν δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου που ασχολούνται με την Ουκρανία θα μεταβούν επιτόπου τον Οκτώβρη για να ελέγξουν τη συμμόρφωση με τους όρους που απομένουν για να εκταμιευτεί η τρίτη δόση. Ρωτήσατε για το χρονοδιάγραμμα και αυτή θα είναι μία αποστολή που θα είναι καθοριστική σημασίας. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημά σας σχετικά με την αντιμετώπιση της διαφθοράς και συναφών μέτρων από τα μέτρα αυτά που σας διάβασα και που εκκρεμούν Κάποια εξ αυτών σχετίζονται με το θέμα της ε, καταπολέμησης της ε, διαφθοράς. Αλλά το γεγονός ότι εκκρεμούν, όπως σας είπα, αυτό ε, σημαίνει η Επιτροπή συνάγει ότι δεν έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα θέματα που θα εξετάσουμε πολύ πιο προσεκτικά και περισσότερο σε βάθος. το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προφανώς και ενημερώνονται με συγκεκριμένο σημείωμα πριν εκταμιευτεί μία δόση για το κατά πόσο πληρούνται οι όροι όχι. Αυτό λοιπόν θα γίνει και τώρα και για την τρίτη δόση. Okay, so, uh, dear colleagues, thank you for this. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και την Επιτροπή που τοποθετήθηκε και απάντησε σε ερωτήσεις. Ολοκληρώσαμε και με το σημείο υπερθμών 9 της τη ε, διάταξης. Ε, το ε, επόμενο θέμα είναι η συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών η ε, βοηθή των ε, συντονιστών επιτρέπεται να είναι παρόντες και κάποιοι νομικοί σύμβουλοι, αλλά τέλος πάντων αυτή η συνεδρία θα λάβει η χώρα στις 11, που σημαίνει ότι έχουμε διάλειμμα 12 λεπτών και θα ξανασυντηθούμε εδώ για τις συνεδρίες των συντονιστών στις 11 ακριβώς. Ευχαριστώ.